Γι' αυτό θα θέλαμε να τις έχουμε μέχρι αύριο το πρωί. Ναι, θα σας απαντήσω τώρα. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έπρεπε να ετοιμάσουν αυτόν τον κατάλογο που τον παρέδωσαν πριν από δύο ώρες. Είναι πολύ ε, πρόσφατος κατάλογος που μόλις ετοίμασαν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Θα σας τον παρουσιάσω δε τώρα αμέσως. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρλο Κασίνη. Πρόεδρε, θα σεβαστούμε τις αποφάσεις σας, αλλά τη στιγμή που υπάρχουν επιφυλά... υπάρχουν επιφυλάξεις για ορισμένες τροπολογίες, ε, δεν σχετίζονται άμεσα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω όμως ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έχει γενικότερες αρμοδιότητες να υποβάλει προτάσεις ως προς την τροποποίηση του κανονισμού. Είτε προταθεί από μεμονωμένους ε, βουλευτές, είτε από ομάδα. Στα πλαίσια λοιπόν μίας ε, ευρύτερης αναθεώρησης του κανονισμού σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας για να γίνουν ορισμένες διορθώσεις δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί απαράδεκτο, αυτές οι τροπολογίες να θεωρηθούν μη αποδεκτές δηλαδή, διότι ορισμένες τροπολογίες μεταφέρουν στον κανονισμό το πνεύμα της ε, Λισαβόνας. Και πολύ συχνά αναφέρονται στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Μιλάμε για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου. Εμείς βεβαίως θα σεβαστούμε τις αποφάσεις σας, αλλά έκανα σκόπιμο να υποβάλω αυτή την παρατήρηση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, ο κύριος Σάντορ Ταμπάτζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση δείχνει σαφώς πως έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μια διαδικασία σημαντική μεταρρυθμίσεων που δεν θα μπορεί να καλυφθεί με μια μοναδική έκθεση. Ευχαριστώ τον, τον κύριο Μάρτιν και τον κύριο Κορμπέτ και όλους τους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που εκκρεμούν που θα πρέπει νομικά να προσδιοριστούν στο μέλλον. θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Με χαρά βλέπω ότι το Κοινοβούλιο δήλωσε σαφώς ότι υποστηρίζει τα θεμελιώδη, το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά ε, έχουν ζητηθεί παρεκκλήσεις από αυτό το χάρτη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα που είναι ανοιχτά, τα οποία δημιουργούν κάποιες ανησυχίες, θέματα που θεωρούνται ότι δεν ανήκουν ακόμα στο κοινοτικό και εκτιμένο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν κυρίως σε ό,τι αφορά τα θεμελιώ... το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να προσδιορίσουμε επακριβώς ποια δικαιώματα θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση. Και το θέμα της γλώσσας στη Σλοβακία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λένε ορισμένοι ότι δεν ενδιαφέρει την Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, ε, έχω έρθει εδώ ως δημοκράτης ως κάποιο που έχει αναλάβει δημοκρατική εντολή. Μια εντολή παρόμοια με εκείνη που έχουν όλοι όσοι εξελέγησαν στο Κοινοβούλιο. Βρίσκομαι μπροστά σας επίσης σαν κάποια που έρχεται από μια χώρα με περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχει πολλά να τονίσει σε ό,τι αφορά εκείνους που προσπαθούν να καταλύσουν, να καταλύσουν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Είχα έρθει λοιπόν με εμπιστοσύνη εδώ, αλλά ως πρώτη φορά νεοεκλογήσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνω ότι αποκλείομαι από τη συναντήσεις των συντονιστών, ότι δεν έχω φωνή στη διάσκεψη των Προέδρων και ότι τα θέματα αυτά αποτελούν ε, αντικείμενο συζητήσεων και πολύ χαίρομαι που ακούω ότι προσπαθείτε να λύσετε όλα αυτά τα θέματα αλλά σας καλώ κύριε Πρόεδρε τα θέματα αυτά να τα ολοκληρώσετε, να τα λύσετε το ταχύτερο δυνατό διότι είναι σημαντικό η δημοκρατική εντολή αυτού του Κοινοβουλίου να γίνει σεβαστή και σας καλώ να συναντήσετε τους ε, μη εντεταγμένους οι οποίοι και αυτοί είναι δημοκράτες και θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το θέμα. Ε, Ο κύριος Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι Μάρτιν, ε, θέλω να συγχαρώ για τα θέματα που περιλαμβάνει η έκθεση για τους στόχους που επιτύχαμε. Πρέπει να σας πούμε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γίνει ένα πλήρες και ισότιμο κοινοβούλιο και έφτασε ε, στην θέση την οποία προέβλεπαν αρχικά οι συνθήκες ε, και η ε, πολιτικές ομάδες και ε, το Προεδρείο και θεωρώ ότι είναι βασική απόφαση ε, των, της διασκέψεως των Προέδρων και των Επιτροπών. Ο, θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να μην συνεργάζονται με πλήρη συνυπευθυνότητα οι εθνικές επιτροπές με τις ευρωπαϊκές επιτροπές. Θεωρώ ότι ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έρχονται οι πρόεδροι και όχι οι αντιπρόεδροι αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και η Ολομέλεια δεν μπορεί να κρίνει εάν είναι σωστές ή λανθασμένες ε, οι αποφάσεις ε, των υπηρεσιών. Θα έπρεπε να αποφασίσει η Ολομέλεια και μόνο έτσι θα μπορέσουν να προστατευθούν οι βουλευτές διότι διαφορετικά δεν μπορώ να δεχθώ να ε, περιορίσουμε τις ε, αρμοδιότητες των Ευρωβουλευτών εδώ. Ευχαριστώ. ο Ρομπέρτο Γουελετιέρη για 1,5 λεπτό. Με την ε, έγκριση της έκθεσης Μάρτιν, στην ουσία ανταποκρινόμαστε σε μία αδύρυτη ανάγκη, δηλαδή να εγκρίνουμε μία έκθεση που θα αποτελέσει συνέχεια, ε, μάλλον θα αποτελέσει εμπροστοφυλακή της συνθήκης της Λισαβόνας. Μιλάμε για μία νομοθετική διαδικασία, μία δημοσιονομική διαδικασία και μία θεσμική εξισορρόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για την αναθεώρηση των συνθήκων και για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων που φέρουν ε, συγκεκριμένη ευθύνη για την ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης ε, νομιμοποίησης και όχι ενός ε, γραφειοκρατικού βραχνά. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν οι τροπολογίες αυτές που σχετίζονται άμεσα με την έκθεση και μετά θα μπορέσουμε να εξετάσουμε την αναθεώρηση του κανονισμού μας εις βάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία ε, αποτελούν αναπόσπαστο έργο της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων και αναφέρομαι στο θέμα της ε, τροπολογίας που αφορά τους παρατηρητές. Θα πρέπει οι παρατηρητές να είναι πρόσωπα που έχουν εκλεγεί ε, μέσα στα πλαίσια των Εθνικών Κοινοβουλίων του Ευρωπαϊκού. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τους εισηγητές, ιδιαίτερα τον κύριο Μάρτιν και βεβαίως τον κύριο Κόρμπετ και να πω σε σχέση με τις τροπολογίες του κανονισμού ότι θα πρέπει να τονίσουμε ένα σημείο που αφορά τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρέει από αυτόν τον κανονισμό και τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία σχετίζεται άμεσα με τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις δύο μορφές νομιμότητας, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία. Αυτή που απορρέει από τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μηχανισμούς ελέγχου, νομοθετικούς μηχανισμούς και από την άλλη πλευρά την ε, δημοκρατική συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών. Γι' αυτό συμφώνω απόλυτα με τις προτάσεις. Δεν συμφωνώ με τον Σάθο Ντάφο, ο οποίος λέει ότι πρέπει να αφήσουμε για αργότερα τους μηχανισμούς συσχετισμού με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να υπάρχουν, πιστεύω, παράλληλα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και δέχομαι τις προτάσεις ιδιαίτερα του κ. Μπρόκ ως προς την εκπροσώπηση της ΚΟΖΑΚ και συμφωνώ με τις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Μπρόκ και άλλων συναδέλφων σε σχέση με την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με άλλες συναφείς υπηρεσίες. Μάριο Μάουρο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Μιλάμε για αλλαγή φύσης και εργασίας των θεσμικών μας οργάνων. Μιλάμε για νομοθετικούς μηχανισμούς που θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ευκαιρίες που μας προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς θα κινηθεί η κοινοτική μηχανή στο εγγύς μέλλον. Γι' αυτό, αυτό που είναι το πραγματικό διακύβευμα είναι η ενίσχυση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα καθώς και του επικουρικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον μας, διότι δεν λάβαμε επαρκώς υπόψη σε αυτή τη φάση τον πολίτη, τον πολίτη υπό την τελεολογική έννοια, διότι η διαδικασία στην οποία φτάσαμε είναι ικανοποιητική, η Ευρώπη πια μετράει για τη ζωή των πολιτών, αλλά αντί να βάλουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της πολιτικής, δυστυχώς έχουμε χειραγωγήσει την επικουρικότητα για να προωθήσουμε τα θεσμικά όργανα και τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είναι αποφασιστική σημασίας. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα εποπτείας για να έχουμε μια πραγματική αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων που εξετάζει το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε σχέση με την τήρηση αυτής της αρχής της επικουρικότητας, που θα πρέπει να είναι σημείο εκκίνησης των θεσμικών οργάνων και όχι να ορίζουν τη ζωή των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ. Μέντες Δεβίγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για το παραδεκτό των ε, τροπολογιών και το κατά πόσο μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Εσείς ε, αναφερθήκατε στον κύριο Καζίνη, δηλαδή σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων. Εμείς είμαστε ένα κυρίαρχο όργανο και μπορούμε να αποφασίσουμε κατά πόσο μια τροπολογία είναι αναγκαία ή όχι. Βρισκόμαστε σε ένα νέο στάδιο εργασιών Γι' αυτό θα ήθελα να, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εξουσίες, ε, με σύνεση βεβαίως, και να κάνετε αυτό που αναμένουμε όλοι από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα παρακαλέσω τον εισηγητή να πάρει το λόγο, κύριε Ντέιβιτ Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στη συζήτηση και θέλω να επανέλθω αυτό που μόλις μας είπε ο κύριος Μέντες Ντεβίγκο. Ο κύριος Κασίνη πολύ σοφά είπε ότι υπάρχουν τροπολογίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Απολύτως καμία σχέση και που θα, θα μπορούσαν να δεχθώ ορισμένες να ψηφιστούν πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε μια χωριστή συζήτηση για το θέμα αυτό προτού περάσουμε στην ψηφοφορία. Θέλω να καταθήσω ωστόσο σαφές. Τίποτα δεν εμποδίζει τα μέλη να υποβάλουν ε, θέματα όπως αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φόξ, αφαίρεση από το Προεδρείο κάποιων εξουσιών υπέρ των κρατών μελών. Δεν έχω καμία αντίρρηση να υποβληθούν σε συζήτηση όλα αυτά τα θέματα στο μέλλον. Αλλά στροπολογίες όπως ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων Μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τη συνθήκη της Αβώνας, αλλά έχει σχέση, όπως είπε ο κύριος Κασίνη, με το πνεύμα της εφαρμογής της συνθήκης της Αβώνας, διότι αλλάζει η σχέση με τις εθνικές, τα εθνικά κοινοβούλια ε, μετά από την ε, έναρξη ισχύω της ε, συνθήκης της Λισαβόνας το θέμα των αντιπροεδριών στις επιτροπές και τα θέματα που έχουν σχέση με τον Προεδρείο δεν είναι θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη συνθήκη της Αβώνας και γι' αυτό δεν πρέπει να μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα σταματήσει η συζήτησή μας και θα κηρύξουμε τη λήξη της απόψινής μας συνεδρίασης.